Yes, friends, uh, we'll start the φίλοι μου, αρχίζει η συνεδρίαση, διότι είναι μακρά η μέρα που μας περιμένει και οι ψηφοφορίες ακόμα μεγαλύτερες και θα πρέπει τώρα έτσι να το προωθήσουμε ε, το όλο θέμα. Ε, πάμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη, τη κανονική. Έχουμε όλες τις γλώσσες στη διάθεσή μας, εκτός από τα μαλτέζικα, τα κροατικά και τα γοηδελικά. Σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη, έγκριση των πρακτικών συνεδρίας 26 Απριλίου. Μπορούμε να τα εγκρίνουμε. η διάταξη αυτή καθ' αυτή. Έχουμε την έξι κυρία Σατζέα για τις κατευθυντήριες γραμμές την απασχόληση. Μετά έχουμε την γνωμοδότηση του κυρίου Σιλικιώτη για τα δημοσιονομικά της Ευρωζώνης. Μετά έχουμε την κυρία Γιασλοβιέκα την έκθεσή της για το πρωτόκολλο Συμφωνία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ελβετίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχουμε ψηφοφορία στη συνέχεια η οποία θα αρχίσει στις 5. Και η σειρά των ψηφοφοριών τώρα θα γίνει ως εξής. Πρώτα, η συμβολή της Επιτροπής έμπλη στο διαρθρωμένο διάλογο. Δεύτερον, η γνωμοδότηση του κ. Πυρίνσκη για την προετοιμασία της μετακλογικής αναθεώρησης του PDP 2014-2020, το στο νομικό πλαίσιο. Μετά θα ψηφίσουμε την έκθεση Benify για τους ε, πρόσφυγες, κοινωνική ένταξη και σωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και τελευταία ε, θα είναι η έκθεση της κυρίας Στεβεν. Πρώτα το 10 λοιπόν και μετά το 9 στην ημερήσια διάταξη για την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ε, είναι μακρά λοιπόν ε, αυτή η ώρα της ψηφοφορίας, αλλά θα αρχίσουμε με τη σειρά με την κανονική μερίσια διάταξη πριν πάμε στις ψηφοφορίες. Ορίστε, ποιος έχει ερώτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω μια διαμαρτυρία. Την περασμένη εβδομάδα, λέει ο κύριος Δομινίκ Μαρτά, και ο πήγα μετά από πρόσκληση του κυρίου Κράσνοπτέρσκι για να συζητήσουμε την ε, σχετική έκθεση ο κύριος συγητής είχε ε, κρατήσει κάποιες από τις δικές μας τροπολογίες για να τις εντάξει στις συμβαστικές. Και πριν καν μελετηθεί ε, η συμβιβαστική τροπολογία, οι σοσιαλιστές, η και το ΕΛΚ εξέφρασαν μια θέση αρχής που έλεγε ως εξής. Ε, αρνούνται κατηγορηματικά πριν διαβάσουν καν τις δικές μας τροπολογίες και τις συμβιβαστικέ, αρνούνται να τις ψηφίσουν σε περίπτωση που μια συμβιβαστική είχε μέσα δική μας τροπολογία. Ε, διαμαρτύρομαι εντόνως. Ε, αυτή η θέση αρχής και αντιδημοκρατική είναι και το θέμα δεν είναι να συνεχίσουμε την προεκλογική μας εκστρατεία όταν είμαστε σε συνεδρία οδών εισηγητών, αλλά να υπερασπιστούμε όσο γίνεται καλύτερα το συμφέρον του συνόλου των Ευρωπαίων συμπολιτών μα. Σας λέω λοιπόν και δημοσίω ότι θα αποσταλεί επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής μα Ευχαριστώ. This is a point of Αυτό είναι διαδικαστικό. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Κάζα. Thank Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δικαίωμά μα είναι να το κάνουμε. Δυστυχώ η η ε, ε, Ένωση ε, για την Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας έχει κάποιες θέσεις που είναι απέναντι τελείως ε, και κατά μέτωπο ε, διαφωνούμε. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Έχει να κάνει με τις ιδέες και την ιδεολογία του κόμματός του, με το οποίο δεν συμφωνούμε και δεν συνεργαζόμαστε. Thank you. Ευχαριστώ. Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόληση των κρατών μελών. Δίνω το λόγο στην κυρία Ατζέα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Εγώ, παρότι λυπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο Χέγγελ που μου έδωσε τη δυνατότητα να ε, ε, αναλάβω αυτήν την έκθεση και να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις ε, για την ε, συνεργασία τους. Την προηγούμενη χρονιά το Κοινοβούλιο εκλήθη να λάβει θέση πάνω σε μια απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές ε, υπέρ της απασχόλησης. Η πρόταση του Συμβουλίου, έτσι όπως μας είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Απασχόλησης, ε, ήταν απλώς μια δήλωση προθέσεων. Βεβαίως ε, ανέφερε μεγαλύτερη δέσμευση όσον αφορά την απασχόληση, ε, απασχόληση παρόλα αυτά παρέμενε απολύτως ασαφής όσον αφορά τα συγκεκριμένα απτά και πρακτικά μέτρα τα οποία ήταν απαραίτητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την μεγάλη ε, και διάχυτη ένδια καθώς επίσης ε, και την ε, έλλειψη απασχόλησης. Δεν δίνονται συγκεκριμένα τα στοιχεία όσον αφορά είτε τη φτώχεια είτε την απασχόληση. Δεν ξέρω, εμείς είχαμε εδώ ασχοληθεί με το θέμα αυτό, γιατί δηλαδή δεν είχαν συμπεριληφθεί συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά την, τα συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη ιδέα Επομένως έπρεπε να ε, βελτιωθεί η πρόταση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εντάξαμε συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά και τη φτώχεια και την απασχόληση και κάναμε συγκεκριμένες και πολύ δυνατές προτάσεις. Η πρόθεσή μας ήταν ακριβώς ε, να ε, ε, κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση έτσι ώστε με συγκεκριμένο τρόπο να γίνουμε αποτελεσματικοί. Είχαμε υπευλήσει ανθρωπολογίες οι οποίες μετά έγιναν συμβιβαστικέ λύσει και γι' αυτό ακριβώ, μέσω μάλλον αυτών, μπορέσαμε να εισάγουμε συγκεκριμένα πράγματα όπω α πούμε η κοινωνική προστασία, όπως είναι η προστασία ναι, των ανέργων αλλά και η επανένταξή του, ειδικά των μακροχρονίων ανέργων. η Η γραφειοκρατία που είναι ιδιαίτερο άχθος για τις μικρές κυρίως και μεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό λοιπόν εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να ελαφρυνθεί αυτό το δημοσιονομικό διορθώνο, το γραφειοκρατικό άχθος ε, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για τους αυτοαπασχολούμενους ε, έτσι ε, επίσης μέτρα έτσι ώστε η παράνομη γκρίζα εργασία ε, να αντιμετωπιστεί. Είχαμε μάλιστα και διοργάνωση μιας ακρόασης για την πλατφόρμα της γκρίζας και αφανούς εργασίας. Επίσης, ε, κάναμε συγκεκριμένες προτάσει όσον αφορά την συνεταιριστική οικονομία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, δούμε μια καινούρια κατάσταση, ε, γιατί βλέπουμε, α πούμε, με, την με το τρίτο μνημόνιο στην Ελλάδα έχουν, γίνει, έχουν ληφθεί μέτρα πολύ συγκεκριμένα όσον αφορά τις, τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά που είναι πάρα πολύ βαριά, είναι μια μεταρρύθμιση εξαιρετικά βαριά. Ε, η εξαιρετική εργασία της ε, Επιτροπής ε, στην ουσία όμως αγνοήθηκε από το Συμβούλιο. Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο το Συμβούλιο ξαναζητά από το Κοινοβούλιο να δεχτεί εκείνη την πρώτη πρόταση που είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Απασχόλησης και που η Επιτροπή Απασχόλησης την είχε κρίνει ασαφή και χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους συναδέλφους ε, γιατί υποστήριξαν ότι πρέπει να εργαστούμε ακόμα περισσότερο στον αφορά το έγγραφο αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη τη στάση του Συμβουλίου, εγώ προσπάθησα να βασίσω την εργασία αυτή τη ε, χρονιά σα σε τούτη την έκθεση και ε, επομένως ε, και οι προτάσει οι οποίε που κάνω και αυτή τη χρονιά ήδη έχουν ενταχθεί στην προηγούμενη έκθεση και τις έχουν συμμεριστεί οι συνάδελφοι που είχαν δουλέψει και στην προηγούμενη έκθεση. Θεωρώ ότι η υποχρέωσή μου είναι με μετεπιτάσεως να επαναλάβω αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει πριν από ένα χρόνο στην Επιτροπή μας και τον προηγούμενο Ιούλιο στο ε, στο, στην Ολομέλεια. Ε, εξακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ενιαία, κοινή ε, και ενωτική θέση, την οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβει υπόψη του το Συμβούλιο. Έχω υποβάλει επίσης σειρά τροπολογιών που κυκλοφόρησαν μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, με τρόπο ώστε για μία ακόμα φορά να έχουμε την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την σημασία της εργασίας μας και όχι να δουλεύουμε μήνες και μήνες πάνω σε ένα έγγραφο ε, το οποίο όπως την προηγούμενη χρονιά θα αγνοηθεί πλήρως από το Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν και από αυτή την οπτική γωνία εγώ είμαι απολύτως διατεθειμένη ε, να συνεργαστώ με τους Κιώδης, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία ε, την οποία θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αντιπρόεδρε Γιάννη Βιέτσκα, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά Λάουρα προσωπικά για την ε, προετοιμασία αυτού του σχεδίου έκθεσης και νομίζω ότι αναφέρει στα σημαντικότερα πράγματα. Πρώτον, οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δημοσιεύτηκαν το 2015 δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη από το Συμβούλιο. Πιστεύω ωστόσο ότι αν θέλουμε να αξιολογήσουμε τις εργασίες του Συμβουλίου, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς καλύτερα. Νομίζω, για παράδειγμα, ότι οι συστάσεις μας θα πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές. Θα πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένες προτεραιότητες και όχι να κάνουμε έναν κατάλογο επιθυμιών. Γιατί έτσι θα καταστήσουμε τις συστάσεις μας αυτές και πιο ε, κατανοητές. Ξέρω, δεν είναι εύκολο αυτό το έργο. Θα πρέπει να υπάρξει συμβασμός μεταξύ των πολιτικών ομάδων και υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικές απόψεις, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε το έργο μας να είναι στοχευμένο και στόχοθετημένο. Να ώρα να ε, μιλήσω για αυτό που προτείνονται εδώ. Το ζήτημα που συζητούμε είναι ότι οι συστάσεις αναχώρα θα πρέπει να έχουν ένα διαφοροποιημένο περιεχόμενο, σημείο 4, και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για αυτά που πρότεινε η κυρία Σοφία Ριμπέιρο. Θα πρέπει να μιλήσουμε ως Επιτροπή Απασχόλησης για τρεις δείκτες συγκεκριμένα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για, για τρεις πυλώνες. Μακροχρόνια ανεργία, ανεργία μεταξύ των νέων, Αυτά πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη στις συστάσεις μας. Και εκ μέρου του ΕΛΚ θα ήθελα να μιλήσω και για την τροπολογία 5. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι οι πολιτικές λιτότητας που ακολουθήθηκαν σε κάποιες χώρες ε, ε, ευθύνονται για την αύξηση της ανεργία. Ήταν απαραίτητα τα μέτρα λιτότητα. Ενδεχομένω να μην εφαρμόστηκαν σωστά ή να εφαρμόστηκαν για υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Και αυτό έχει ως συνέπεια να πληγεί η οικονομία και η δυναμική της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας δεν ήταν απαραίτητα. Ήταν. Επίσης, εμείς θέλουμε να υπάρχει μεν αναφορά στην ανάγκη θέσπισης κατώτατου μισθού, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται σεβαστό και το, η αρχή της αναλογικότητας, της επικουρικότητας, με συγχωρείτε. Και θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστούν οι αρχές που είχαν ε, ψηφιστεί το 2015 από το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Χαβι από τους Σοσιαλιστές έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς, η ομάδα μας θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια, τη Λάουρα ε, Ατζέα, για το έργο της θέλουμε να τονίσουμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, τη γνώμη και τη γνωμοδότηση που πρέπει να έχει η Επιτροπή Απασχόληση και το Κοινοβούλιο στι συστάσει του Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη για τι πολιτικέ απασχόλησει. Όπω πολύ ωραία μέχρι τώρα εξηγήσατε. Το 2015 ήταν πλήρης η άγνοια, ε, όσα λέγαμε εμείς για τις τελευταίες συστάσεις του Συμβουλίου. Και αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να επανέλθουν όλε αυτέ οι γνωμοδοτήσει και η προηγούμενη εργασία που υπάρχει από πλευρά τη Επιτροπή μα και να τα συμπεριλάβουμε ξανά και να τα στείλουμε στο Συμβούλιο μήπω και τα λάβουν υπόψη. Τι κάνει λοιπόν η πρόταση αυτή τη νομοδότηση. Συστήνει διάφορα πράγματα που εμείς ε, ε, συμφωνούμε. Ε, επισημαίνει και πάλι στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι από πέρσι τα έχουμε πει αυτά. Ε, υπενθυμίζει τις προκλήσεις που έχουμε απέναντί μας ε, και μπροστά μας την ε, ανισότητα, τη φτώχεια, την απασχόληση και ε, τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους στόχους μας για το έτος 2020 στα κοινωνικά θέματα. Βεβαίω έχει σχέση και με την παιδεία αυτό και με την κατάρτιση και την απασχόληση. Επίσης πολύ ε, καλά κάνει ε, η συγγήτρια που επισημαίνει ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Εμείς κάνουμε εδώ πέρα τόση δουλειά, γνωμοδοτούμε και κατόπιν μας αγνοεί το Συμβούλιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και επίση πρέπει να επιμείνουμε οι κοινωνικοί δείκτε να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με του μακροοικονομικού. Αυτά λοιπόν προτείνει η συγκήτρια. Μας, μας βρίσκουν σύμφωνο στην ομάδα μας, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το συμπληρώσουμε και να το ενισχύσουμε σε διάλογο που θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες. Να υπόψη τα όσα ήδη έχουν εγκριθεί, όπως είπε και η σκιώδης ε, του ΕΛΚΑ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα και θα πρέπει να έρθουμε τώρα να τα συμπληρώσουμε με ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανισότητα, με τη μακροχρόνια ανεργία, καθώς επίσης και με την ανεργία των νέων, που είναι τα θέματα που μας ανησυχούν περισσότερο. Thank you. Mr. Bashir is Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασίρ απουσιάζει. Τον εκπροσωπεί κάποιος. Η κυρία Μάκεντάιρ, η CR, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο Σάλς Μπασίρ δυστυχώς, ο οποίος είναι ο σκιώδης, δεν μπόρεσε να είναι εδώ και ζητά συγγνώμη γι' αυτό και διαβάζω αυτά που μου έχει αφήσει. Πρώτα απ' όλα ευχαριστεί την Λάουρα, ε, την εισηγήτρια για την εργασία της. Η ομάδα ECR θέλει να στηρίξει την πρόταση της Επιτροπής έτσι όπως προτείνεται, αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε τόσο πολύ τις προτάσεις της εισηγητρίας ε, για την τροποποίηση ορισμένων σημείων. Ε, εδώ προκύπτει ένα ζήτημα αρμοδιότητας κατά τη δική μας άποψη. Συζητούμε τις κατευθυντήρες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησεις, οι οποίες όμως στο μεγαλύτερο τμήμα τους παραμένουν αρμοδιότητα αποκλειστικά των κρατών μελών Επομένως λοιπόν δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε να ξανανοίξει η συζήτηση για τις κατευθυντήριες γραμμές επί των οποίων έχουν ήδη συμφωνήσει τα κράτη-μέλη. Επίσης αμφισβητούμε κατά το πόσο αυτό είναι ο τρόπος να ακουστεί καλύτερα η φωνή μας στην Επιτροπή Απασχόλησης. Υπάρχουν ε, σημεία επί των οποίων το Κοινοβούλιο έχει συναπόφαση. Επιπροσθέτως, έχουμε ε, υποβάλει και πολλές, πολλές εκθέσεις ε, πρωτοβουλίας ε, που καταδεικνύουν τη θέση του Κοινοβουλίου επί σειρά θεμάτων. Επί θεμάτων. υπάρχουν πολλά στοιχεία και πολλοί τομείς επί των οποίων μπορεί πραγματικά να έχει σημασία να ακουστεί η φωνή της Επιτροπής μας και όχι πάνω σε ήδη συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν είναι κανείς εδώ από τους φιλελεύθερους. Κανείς από την ΚΟΕ. Κανείς από τους πράσινους επίσης. Οπότε ο κύριος Μαρτάν από το ΙΕΝΕΦ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ομολογώ ότι ε, είμαι λίγο προβληματισμένος ε, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάτε. Μιλάτε για τροπολογίες τις οποίες ενδεχομένω έχει προετοιμάσει η κυρία Ατζέα, αλλά εγώ δεν τις γνωρίζω, δεν μου έχουν γνωστοποιηθεί αυτές οι τροπολογίες, άρα δεν καταλαβαίνω ε, τι συμβαίνει. Αντιθέτως, ε, αντιθέτως λέω. Ίσως ε, θα μπορούσε να μου εξηγήσει η κυρία Τζέα γιατί φέρθηκε έτσι απέναντί μας. Πάντως ακούγοντά σας ε, λέτε ότι το Συμβούλιο και, το και η Κομισιόν δεν, σας, δεν μας λαμβάνουν υπόψη και άρα δεν χρησιμεύουμε σε τίποτα. Κάπου αυτό με ευχαριστεί και με ικανοποιεί πρέπει να σας πω. Κατανοείτε ότι αυτό το κοινοβούλιο είναι οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς αλλά όχι δημοκρατικό. Δηλαδή ένα, ε, ένα κοινοβούλιο το οποίο μπορεί να συζητά και να συνδιαλέγεται και μετά το Συμβούλιο αποφασίζει και λέει «Α, αυτό που αποφασίσατε εμείς δεν το αποδεχόμαστε». Ε, οι κατευθυντήριες γραμμές ε, για την απασχόληση υφίστανται εδώ και χρόνια και εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι δεν έχει υπάρξει καμία τροποποίηση. Βλέπουμε ότι οτιδήποτε είναι επιβλαβές ή επιζήμιο για την απασχόληση, μετανάστευση, ενσωμάτωση των προσφύγων δια της εργασίας, κινητικότητα εργαζομένων, ε, η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, όλα αυτά τα οποία δυσαρεστούν τις χώρες ε, και που δημιουργούν πρόβλημα στην απασχόληση των ε, δικών μας πολιτών δεν έχουν αλλάξει. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο λέει και εξηγούν ότι εάν όλα αυτά δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούν επειδή δεν υπάρχει αρκετή Ευρώπη. Εγώ ε, συμμερίζομαι μαζί σας ε, την αίσθηση απασχόλησης ε, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα... και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και εσείς να ανοίξετε τα μάτια σας. Κύριε Μαρτάν, μπορείτε να μας... Νομίζω ότι οι τροπολογίες ήταν δημόσιες και μπορούσατε να τις είχετε διαβάσει και εσείς και όλοι βεβαίως. 6 Ιουνίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. 7, με συγχωρείτε. 7 Ιουνίου. Άρα όσοι δεν είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις τροποποίησης της πρότασης αυτής. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει 21 Ιουνίου και στις 13 και 14 Ιουλίου θα γίνει ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή απασχόληση. Σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Δημοσιονομική εικονότητα της Ευρωζώνης και επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τη συμπληρωματικότητα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο κύριος Σιλικιώτης δεν είναι εδώ. τον αντικαθιστά όμως ο συνάδελφος, παρακαλώ συστηθείτε για να μας πείτε ποιος είστε παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Sí. <laughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους του συντρόφου Νεοκλή Σιλικιώτη. Θα παρουσιάσω λοιπόν τις δικές του θέσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θα, στα, θα σας τα διαβάσω, αυτά που μου έστειλε εκείνος. Και θα το κάνω στα αγγλικά. Ελπίζω να μην είναι υπερβολικά έντονη η πορτογαλική μου προφορά στα αγγλικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία μου σήμερα και ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς για την κατανόησή σας αλλά και τους, τον συνάδελφό μου που με αντικαθιστά σε αυτή την πρώτη εξέταση της γνωμοδότησης για τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Ο λόγος της απουσίας μου είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο, έπειτα από τις εκλογές που διεξήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τον προβληματισμό και τις σκέψεις που θα εκφράσετε εδώ και σας διαβεβαιώ ότι αναπομονώ και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία μαζί σας. το γενικό σκεπτικό πίσω από αυτή την γνωμοδότηση ήταν να δώσουμε έμφαση σε, στην κοινωνική διάσταση της δημοσιονομικής οικονομικής χωρίς να μπούμε σε οικονομικές λεπτομέρειες. Αυτά μπορούν να τα κάνουν οι Επιτροπές ε, Προϋπολογισμών και Οικονομικών και Νομισματικών ε, Υποθέσεων. Ταυτόχρονα εξετάζουμε το γεγονός ότι τα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα εντείνονται. Πλήγματα στα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Ιστορικά υψηλή ανεργία μεταξύ των νέων. Υπάρχει πλέον, ζούμε μια, σε μια ένωση πολλών ταχυτό, ταχυτήτων όπου πλήττεται σοβαρά η κοινωνική συνοχή. Αυτές είναι και οι σκέψεις που οδήγησαν στη σύνταξη της πρώτης παραγράφου, όπου γίνεται έκκληση να δημιουργηθούν νέες αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης, να ενισχυθεί η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και να γίνεται πλήρως σεβαστή η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παράγραφοι 2 και 3 βασίζονται στο ίδιο πνεύμα. Πολλές δυνάμεις σε αυτό το κοινοβούλιο τη αριστερά θεωρούν ότι η οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης είναι μονόπλευρη. Γι' αυτό και τονίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αγνοεί τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές ε, λιτότητας που οδηγούν τους πολίτες στην ένδια, αυξάνουν την ανεργία και αυξάνουν τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι άνεργοι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας από 37,5 το 2005 πήγαν στο, 46,9 το 2014 με τάση αυξανόμενη. Η Κομισιόν διακηρύσει, η Επιτροπή μάλλον καλεί να ε, δημιουργηθεί μια, ένας κοινωνικός πυλώνας ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο καλούμε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιδόματος ανεργίας ως τμήμα του κοινωνικού αυτού πυλώνα. Και εμείς δεν συζητούμε την ε, μορφή αυτού του συστήματος εφόσον δεν έχει κατατεθεί ακόμα πρόταση στο Κοινοβούλιο. Λέμε όμως ότι κάθε τέτοιο σύστημα, κάθε μορφή τέτοιου συστήματος θα πρέπει να ενισχύει τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και δεν θα πρέπει να ε, βασίζεται σε όρους διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη που χρειάστηκε, που αναγκάστηκαν να ε, εφαρμόσουν μνημόνια εφάρμοσαν μέτρα χωρίς δημοκρατική λογοδοσία τα οποία ήταν καταστροφικά για τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες αυτές. Στην παράγραφο 5 πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα και τονίζουμε ότι κάθε τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να καταπολεμά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι κάθε επίδομα ε, ανεργίας, κάθε σύστημα επιδόματος ανεργίας δεν θα ε, πρέπει να, αντικαθιστά τις πολιτικές επαναβιομηχάνησης και την ανάγκη να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς θέσεις εργασίας. Με αυτές τις σκέψεις προσβλέπω στα σχόλια και τις παρατηρήσεις των ε, συναδέλφων μου και περιμένουμε να έχουμε μια καλή και γόνιμη συνεργασία. Σε, ε, ευχαριστώ κύριε Πιμέτα Λόπες. Η κυρία Λόπε Φοντανιέ είναι η πρώτη σκιώδης, την οποία όμως αντικαθιστά η κυρία Ριμπέρ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Συνάδελφο Βερόνικα Λόρπε Φοντανιέ κολλείεται και μου ζήτησε να διαβάσω τη δική της γραπτή δήλωση και να σας παρουσιάσει τη θέση τη. Και αρχίζω να παραθέτω. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σιλικιώτη για το σχέδιο έκθεσης και δηλώνω την πλήρη προθυμία μας να συνεργαστούμε μαζί του και με τους υπολείπους για να καταλήξουμε στις συμφωνίες. Η οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει να φαίνεται στους πολίτες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σημαίνει επένδυση ε, στον κόσμο που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση. Η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η απασχόληση, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το δημοσιονομικό έλεγχο. Τούτων λεχτέντων και με κάποιες αλλαγές θα μπορούσα να συμφωνήσω με τις παραγράφους 1 και 6. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ο δημοσιονομικός έλεγχος χρειάζεται για να τονώσει την ανάπτυξη και να δημιουργεί εργασία και απασχόληση βιώσιμη και αηφόρο. Γι' αυτό διαφωνώ με την παράγραφο 3. Ε, ε, μια άλλη υπόθεση που είναι επίμαχη είναι ε, η ασφάλιση του επιδόματος ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να χρειάζεται για τις ασύμετρες ε, αναταράξει και κραδασμού, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι το σωστό εργαλείο εδώ. Στην παράγραφο 4 μπορώ να υποστηρίξω εκείνα που λέει ο συγγητής, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει και στην κοινωνική διάσταση, αλλά όχι με τον τρόπο που εκείνο ζητάει. Ισορροπία με τον οικονομικό πυλώνα, θα κάνω κάποιες απολογίες σχετικά. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω να μου εξηγήσει ο εισηγητής τι ακριβώς θέλει να πει στην παράγραφο 5 ότι δεν συνδέει οικονομική αιρεσιμότητα με τα επιδόματα ανεργία στα κράτη-μέλη. Και πάλι τον ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί του τις επόμενες εβδομάδες. Τέλος της παράθεσης της κυρίας Λόπε Φονταγιά. Ευχαριστώ κυρία Ριμπέρο. Η Μαρία Ζωάου Ροντρίγκης έχει το λόγο. Παρακαλώ σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση ε, και οι συνέλφοι της ε, ΕΚΟΝ συζητούν ε, συμπτωματικά ακριβώς για το ίδιο θέμα του τη στιγμή. Είναι σημαντικό που ασχολείται και εμπλέκεται στη συζήτηση και η Επιτροπή μας. Εδώ παίζεται το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, της Ευρωζώνης, η οποία αντιμετωπίζει ε, πολλαπλά προβλήματα εσωτερικά και εξωτερικά. Έχουν υπάρξει αποκλήσεις όσον αφορά την απασχόληση, όσον αφορά τα ποσοστά, ε, κυρίως όσον αφορά δε τα ποσοστά ανεργίας των νέων. Ε, επίσης ε, υπάρχουν ε, και φθήνουσες πορείες των κοινωνικών προτύπων στις διάφορες χώρες και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε με τρόπο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση και γρηγορότερη ανάκαμψη. Βεβαίως οι προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν και από κάθε χώρα μέλος. Όταν εγκρίναμε την έκθεσή μας όσον αφορά την ετήσια ε, επισκόπηση ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, αλλά οι σωστές ε, μεταρρυθμίσεις και οπωσδήποτε και ε, να υπάρξουν καλές επενδύσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε και το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχία στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πλέον να έχουμε την δυνατότητα να καλύπτουμε τα κενά κενά τα οποία δεν μπορούν πλέον να καλύψουν ε, τα κράτη από μόνα τους. Ε, γι' αυτό λοιπόν και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ έχουν ε, συζητηθεί τα θέματα αυτά και έχουν αναφερθεί πολλά είδη δημοσιονομικής ικανότητας. Δύο είναι τα κυριότερα. Το ένα είναι αυτό που θα βοηθήσει την ανάπτυξη ανάκαμψη και ένα άλλο αυτό το οποίο θα προστατέψει τις χώρες από τα διάφορα σοκ και θα μπορούσε να αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο μία ε, διασφάλιση της απασχόλησης ε, στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Οικονομική Επιτροπή έχουν ήδη συζητήσει και συμφωνήσει για τα δύο αυτά εργαλεία αλλά βεβαίως θα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεράσουν και αυτό το ευαίσθητο θέμα της αρεσιμότητας υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις. Εγώ μπορώ να σας πω ποια είναι η θέση στην ομάδα μου. Εμάς δεν μας απασχολεί η αιρεσιμότητα. Εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι ότι το περιεχόμενο της αιρεσιμότητας ευθυγραμμίζεται με την πραγματική ανάκαμψη και την πραγματική μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση να αφορούν ε, την εκπαίδευση, την καινοτομία, ε, την, ε, τα κοινωνικά οπλοστάσια με τα οποία θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες και βεβαίως η προώθηση των σωστών επενδύσεων. Αυτή είναι η θέση μας λοιπόν όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τούτη τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Τρεβέσιος έχει το λόγο από την ΕΣΕ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ απορρίπτω ε, την ιδέα κοινού προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωζώνη. Για ποιο λόγο θέλει η Ευρωζώνη κοινό προϋπολογισμό. Η απάντηση είναι σαφή. Δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα του ευρώ και τώρα χρειάζεται κάποια μεταφορά πιστώσεων και συμψηφισμός μεταξύ των κρατών μελών. Οικονομική καταστροφή έχει προκαλέσει εδώ και χρόνια το ευρώ. Ε, στην αρχή είχαμε μεταφορά πιστώσεων από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια σε μια φούσκα οικοδομική με κακές επενδύσεις και κακές επιλογές. Συνέπεια, εμείς στη Γερμανία ε, Είχαμε την ε, μαζική ανεργία και την Ατζέντα 2010. Αυτή η φούσκα λοιπόν στο Νότο έσκασε κάποια στιγμή και ήρθαμε να διαπιστώσουμε ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει ε, η οικοδομή ε, τα όσα χάνονται από το ευρώ και την καταστροφή στη βιομηχανία. Είναι κακή η συγκεντρωτική πολιτική. Δεν έχουμε καταλάβει πώς ε, χρειάζεται ένα σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών για να εξισορροπεί και να απορροφά τους κραδασμούς. Το ευρώ λοιπόν είναι ένα ε, στρεβλό κατασκεύασμα, ένα εξάβλωμα από την κατασκευή του ε, και αντί να ομολογούμε τα λάθη μας τώρα προσπαθούμε επανειλημμένα να τα διατρανώνουμε. Τώρα θέλουμε και κοινή οικονομική κυβέρνηση και κοινούς προϋπολογισμούς για την Ευρωζώνη. Εγώ λέω όχι, απορρίπτω το έγγραφο εργασίας. Τα δικά μας έγγραφα εργασία τη Επιτροπής Απασχόλησης πρέπει να λύνουν προβλήματα. Το θέμα είναι πώς ε, θα αποτρέψουμε ε, τα λάθος κίνητρα, τη μεταφορά πιστώσεων από το βορρά στο νότο. Δεν γίνεται με το ευρώ. Οι ε, συνθήκες που έχουν γίνει ε, αντικείμενο διαπραγμάτευση στην Ευρώπη δεν λειτουργούν. Ε, συνεχώς τις παραβιάζουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ρήτρα μη διάσωσης, μη συμμετοχή της ΕΚΤ. Και τώρα ε, ο μηχανισμός ESM ε, πρόκειται να δώσει χρήματα στην Ελλάδα, τη νέα δόση, ενώ απαγορεύεται να συνάπτει δάνεια. Ο Κλέμενς Φούστ διαπίστωσε ότι σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς ε, νομισματικού ταμείου ε, οι Έλληνες πολίτες οφείλουν 87 δισεκατομμύρια στο κράτος τους. Αυτό αντιστοιχεί στο ποσό που έδωσαν οι Γερμανοί φορολογούμενοι για να σώσουν υποτίθεται την Ελλάδα. Και πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στους Γερμανούς πολίτες που έκαναν σκληρές μεταρρυθμίσεις να το αναλάβουν. Ξέρω τι κάνει ο Σόιμπλε, το έχει μεταθέσει το πρόβλημα για το 2018. Η Ιταλία 14 δις ε, μπορεί τώρα επιπλέον να ε, επενδύσει, μάλλον να δαπανίσει ε, και ξεπερνάει όλο το πλαίσιο και η Ισπανία τα αντίστοιχα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την Ευρωζώνη. Δεν ισχύει το δίκαιο, παραβιάζεται κατάφορα συστηματικά και στόχος είναι να διατηρηθεί ένα σαθρό σύστημα. θα πρέπει να επανέλθουν στο κράτος δικαίου οι ε, ενεχόμενοι και οι πρωταγωνιστές. Είναι σκέτη παράνοια αυτό που γίνεται με την Ευρωζώνη. Θα πρέπει να το απορρίψουμε. Το μόνο που ε, αποσκοπεί και στο μόνο ε, που χρησιμεύει είναι να χρηματοδοτούνται προβληματικές δομές. Ε, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί και στη Ιταλία και πάλι δεν κάνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά συγκυριακά ε, κρατικά προγράμματα και νέα χρέη. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στις χώρες αυτές ε, μεταρρυθμίσεις γιατί εκλέγουν εχθρικά προς την Ευρώπη κόμματα. Οι μεταρρυθμίσεις ε, ε, πηγάζουν από κάτω προς τα πάνω και όχι με φυρμάνια και διατάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μικρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ζώνη. Αν θέλουν να πάρουν το δρόμο τους στο καλό Ιταλία και Γάλλοι αλλά όχι με τα λεφτά των άλλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος των φιλελευθέρων στην αίθουσα, ούτε των πρασίνων. Δεν έχει οριστεί σκιώδης από την ομάδα EFDD και έτσι δίνω τον λόγο στην κυρία Μελάν από το ΕΝΕΦ e η οποία επίσης απουσιάζει οπότε φαντάζομαι Ντομινίκ Μαρτάν θα πάρετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή εμείς νομοδοτούμε και μας παρουσιάζουν την Ευρωζώνη ως λύση. Ή τι λύση μάλιστα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Η Ευρωζώνη δεν είναι η λύση, αλλά το πρόβλημα είναι. Και αυτό αποδεικνύει ότι η κρίση δεν είναι συγκυριακή, αλλά διαρθρωτική. Από το ευρώ το ίδιο. Απόδειξη. Η Ευρωζώνη είναι κύριος ο χώρος όπου ε, υπάρχει χαμηλότερη ανάπτυξη από ολόκληρο τον κόσμο. Μιλάω για τις αναπτυσσόμενες, αναπτυγμένες συγγνώμη, λεγόμενες χώρες. Άρα που σημαίνει ότι η Ευρωζώνη και το ευρώ είναι βαρύδι. Και ε, αντί να γίνει αυτό που προτείνει η Γκουε στην νομοδότηση, που ξέρουμε ότι η βάση τους είναι η κατάργηση όλων των εθνών και ε, ένας άλλος κόσμος, εμείς θεωρούμε τελείως το αντίθετο, ότι για να γλιτώσουμε χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, όπως παλιά, η Ευρώπη των πατρίδων, η Ευρώπη των εθνών. Και αν κάθε ένα από αυτά τα κράτη, τα έθνη κράτη είναι ισχυρό, τότε θα είναι ισχυρή και η Ευρώπη. Εσείς τι θέλετε, ε, με, με δύσχυρες χώρες να κάνετε μια ισχυρή Ευρώπη, που είναι αρκετά ανόητο αυτό. Και το αντίθετο αυτό που προτείνεται, ενιαία κυβέρνηση, ενιαίο νόμισμα, ενιαίοι προλογισμοί. Εμείς το, το θέλουμε, βεβαίω δημοσιονομική κυριαρχία, ε, νόμισματική κυριαρχία και επίσης οικονομική και χρηματοπιστωτική κυριαρχία και νομοθετική κυριαρχία. Πράγμα που έχει στο παρελθόν αποδείξει την αποτελεσματικότητά του. Οπότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ ότι βρισκόμαστε τελείως απέναντι και σε πλήρη διαφωνία με τα σχέδιά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούστερ έχει, έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εκείνοι που θέλουν να αναπτύξουν την εσωτερική αγορά ως ουσιαστική βάση της ευημερίας στην Ευρώπη δεν μπορεί παρά να επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη της ε, Ευρωζώνης. Και γι' αυτό το λόγο συζητούμε δικαίως αυτό το θέμα. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από ένα αυστηρό σύστημα, από ένα σύστημα με αυστηρούς κανόνες που δεν λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα εντός της, ε, της ε, Ευρωζώνης. Χρειαζόμαστε ένα πολιτικό σύστημα με πλήρη δημοκρατική λογοδοσία και από αυτή την άποψη χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες προσπάθειες ε, για την ενίσχυση της ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Τι είναι η βασική πρόκληση. Και όλη αυτή η παραφιλολογία ότι το ευρώ ευθύνεται για όλα μας τα δεινά, θα έλεγα εγώ ότι θα ήταν καλό όσοι τα λένε αυτά να ξανακοιτάξουν λίγο την ιστορία και να θυμηθούν πώς και για ποιο λόγο οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του κοινού νομίσματος. Εκεί όπου έχω όμως μια διαφορετική άποψη είναι ε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιδόματος Ανεργίας και τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα τέτοιο σύστημα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κατάλληλο το μέσο αυτό ως οικονομικός σταθεροποιητής. Για διάφορους λόγους. Πρώτον, στον τομέα της ανεργίας δεν έχουμε να κάνουμε με διαρθρωτικό δομικό ε, πρόβλημα αλλά, ε, με συγχωρείτε, συγκυριακό πρόβλημα, αλλά με ένα δομικό πρόβλημα. Και όταν κανείς θέλει να καταπολεμήσει τη δομική ανεργία, τη μακροχρόνια ανεργία, πρέπει να ε, ε ενισχύσει την απασχόληση. Και κατά συνέπεια θα πρέπει η δημοσιονομική πολιτική να επικεντρώνεται στην προώθηση των επενδύσεων σε δυναμικούς ε, τομείς και νομίζουμε ότι το εύση είναι μια καλή αρχή Ωστόσο θα πρέπει από ευρωπαϊκής πλευράς να διωθεί ε, μεγαλύτερη δυνατότητα ε, πραγματοποίησης δημόσιων επενδύσεων στην καινοτομία ιδίως. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα όσον αφορά την, τη μορφή του συστήματος επιδόματος Ανεργία. Αναφέρθηκε βέβαια ότι μια τέτοια μορφή δεν έχει ακόμα προταθεί. Ωστόσο, όποιο ε, σκέφτεται ε, ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ε, και τα εθνικά αντίστοιχα συστήματα και την εναρμόνισή τους, ιδίως ως προς τις βασικές αρχές που τα διέπουν. Αυτή η δουλειά, αυτό το έργο το καθήκον είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι τόσο δύσκολο που ε, με οδηγεί εμένα στο συμπέρασμα ότι ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα επιδόματο ανεργία, αλλά να ενισχυθούν οι δυνατότητε επενδύσεων. Ευχαριστώ, λέει η Προεδρεύουσα. Η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι ε, η 3η Ιουνίου. Η έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης θα γίνει στις 13 Ιουλίου. Η ε, ψηφοφορίες στις Επιτροπές Προϋπολογισμών και Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, που είναι οι καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές, θα γίνουν στις 5 Σεπτεμβρίου, μετά την ε, θερινή διακοπή. Προχωρούμε στο σημείο 6 της σα διάταξης. Πρόκειται για την ε, συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Ντανούτα για Σόφισκα. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα αυτό της σύναψης πρωτοκόλου σχετικά με την ε, προσχώρηση της ε, Κροατίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντίστοιχη ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της χώρας αυτής, εγώ προτείνω την, να δώσει το Κοινοβούλιο τη συγκατάθεσή του. Θεωρούμε ε, ε, ε, διότι είναι απαραίτητη η συγκατάθεση αυτή προκειμένου να μπορέσει να κυρωθεί το πρωτόκολλο αυτό. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά ε, που διευρύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτού σας παρουσιάσω την ε, έκθεσή μου, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, η συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών υπεγράφει το έτος 2000. Επρόκειτο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τότε αποτελούνταν από 15 κράτη-μέλη. Στη συνέχεια, το 2004 και το 2009, η συμφωνία αυτή επεκτάθηκε με το πρωτόκολλο 1 και το πρωτόκολλο 2 αντίστοιχα. Δίνοντας στους πολίτες των ε, κρατών μελών της Ένωσης να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εργάζονται και να διαμένουν στην επικράτεια των άλλων συμβαλωμένων μερών της Συμφωνίας. Έπειτα λοιπόν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σχεδιαστεί να υπογραφεί και ένα τρίτο πρωτόκολλο στην συνθήκη αυτή. Ωστόσο, έπειτα από το δημοψήφισμα που έγινε το 2014, το Φεβρουάριο του 2014 στην Ελβετία σχετικά με την μαζική είσοδο μεταναστών, υπήρξε μια διακοπή ως προς τη σύνταξη αυτών αυτού του πρωτοκόλου. Έπειτα, τον Μάρτιο του 2016, ωστόσο, υπήρξε συμφωνία με την Ελβετία σύμφωνα με την οποία η συμφωνία θα επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει και την Κροατία. Το άρθρο 121 της, ε, του συντάγματος της Ελβετίας δεν είναι συμβατό με τη συμφωνία. Διότι η Ελβετία ζητεί αυτή τη στιγμή οι ελβετικές επιχειρήσεις να έχουν το δικαίωμα να προτιμούν ελβετούς πολίτες ως εργαζόμενους. Ωστόσο, οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις στη βάση της υπηκότητας ενός ε, ανθρώπου στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι το άρθρο 121 του συντάγματος της Ελβετίας δεν είναι συμβατό με τη συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν συμφωνεί και ότι ζητεί την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις επί του θέματος αυτού. Ωστόσο, η δική μου έκθεση δεν αφορά τις λύσεις που αναζητούνται σε αυτό το θέμα. Αντιθέτως, το μοναδικό θέμα της δικής μου έκθεσης είναι η επέκταση της συμφωνίας προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται εφ' και η Κροατία. Και εγώ ως εισηγήτρια προτείνω το Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του στην επέκταση της συμφωνίας. Θεωρώ ότι θα πρόκειται για μια εποφελή εξέλιξη τόσο για την Ελβετία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το εξωτερικό εμπόριο, αλλά και για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο συμβαλωμένων μερών. Το πρωτόκολλο αναφέρει ότι ε, επτά χρόνια έπειτα από τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί πλέον όσον αφορά την αμοιβή ή την ε, προτίμηση εργοδοτών ε, απέναντι στους πολίτες που προσλαμβάνουν. Και για, τον... για να γίνει αυτό θα πρέπει ωστόσο να δώσει επίσης τη σύμφωνη γνώμη του και μια μεικτή επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη που θα έχουν ορίσει αφενός η Ελβετία και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Κροάτες πολίτες που θα θέλουν αυτό το διάστημα, αυτά τα 7 χρόνια να εργαστούν στην Ελβετία θα, θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αφενός θα υπάρχουν οι εργαζόμενοι που θα έχουν άδεια παραμονής από 4 έως 12 μήνες και εκείνοι που θα έχουν άδεια παραμονής άνω του ενός έτους. Σταδιακά οι περιορισμοί αυτοί θα έρονται. Αντίστοιχα μέτρα θα πρέπει να λάβει και η Κροατία στη δική της επικράτεια για τους Ελβετούς πολίτες. Και υπάρχει ρήτρα η οποία αναφέρει ότι μετά το πέρας αυτών των 7 χρόνων η Ελβετία θα διατηρήσει το δικαίωμα να, να ε, εφαρμόζει για άλλα τρία χρόνια μια ρήτρα προστασίας απέναντι στους Κροάτες πολίτες. Με άλλα λόγια, η Ελβετία για δέκα ολόκληρα χρόνια θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει την αγορά εργασίας της από τους Κροάτες. Αυτός ο όρος έγινε αποδεκτός από την ε, κυβέρνηση της ε, Κροατίας και έτσι λοιπόν για όλους τους λόγους που ανέφερα εγώ προτείνω την υπογραφή του πρωτοκόλου 3. Ελπίζω στη δική σας υποστήριξη. Βεβαίως όμως, αν έχετε κάτι να παρατηρήσετε ή να συζητήσετε μαζί μου, είμαι ανοιχτή για ό,τι θέλετε να μου πείτε. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Mr. Κύριος Πυρίνσκι. Yeah, Mr. Πυρίνσκι, the floor Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο στην παρέμβασή μου. Θα ήθελα απλώ να πω εξ ονόματο τη κυρία Στάινροκ, που είναι η δική μα η Ιδρύα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θέλω να εκφράσω τη συμφωνία μας με το σχέδιο έκθεσης κυρίας Γιαζοβιέτσκα. Σας ευχαριστώ. Uh, Έχετε το λόγο. Ε, εισηγήτρια, ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση. Εγώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους της. Και προς εκπροσώπους του Συμβουλίου. Τα τελευταία χρόνια κάποιες χώρες έχουν γίνει μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθούν να έχουμε μεταβατικές περιόδους και προθεσμίες. Δεκαετής ήταν αυτή για την αγορά εργασίας η περίοδος. Εδώ μιλάμε για ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που θέλουμε να την εμβαθύνουμε. Και εδώ πρόκειται για ένα νέο κράτος μέλος με τόσο μακρά μεταβατική περίοδο. Για ποιο λόγο ε, να είναι τόσο μακρά. Ο κύριος Μπέντερ είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να μας διαφωτίσετε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Φοβούμαι ότι δεν μπορώ να σας διαφωτίσω. Για ποιο λόγο ε, η μεταβατική περίοδος είναι τόσο μακρά, προκειμένου ή γενικότερα. Γιατί σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις περισσότερες χώρες έχει θετική επίπτωση στην εγχώρια αγορά εργασίας ο κανόνας των 5 συν 2 ετών ε, έβρισκε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από κάθε διεύρυνση, παγίως δηλαδή. Είναι μια παλιά πρακτική, η οποία συνεχίζεται και για την ε, ε, λόγω υπόθεση το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελβετία. Απλώς μεταφέρεται κάτι που είχε εφαρμοστεί δεν ήταν εσκεμμένη αυτή η ενέργεια, ούτε ε, ε, ζήτησαν ούτε η Ελβετία ούτε το εν λόγω κράτος μέλος να εξαιρεθούν ή να υπάρξει άλλη ρύθμιση. Και εμείς χαιρετίζουμε την υπογραφή από πλευρα των Ελβετών το Μάρτιο του πρωτοκόλου και όπως είπατε και εσείς κυρία ε, εισηγητρία, το Κοινοβούλιο μάλλον θα δώσει τη συγκατάθεσή του στη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Εισηγήτρια, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αυτή. Ωραία. Τέλος. Το χρονοδιάγραμμα είπαμε έως ε, εξής. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών Μαΐου. Αύριο συγκεκριμένα. Και στην Επιτροπή μας θα ψηφιστεί στις 21 Ιουνίου, ενώ αναμένεται να πάει στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο μετά τις θερινές διακοπές. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εδώ την ημερήσια διάταξη και φτάσαμε στις ψηφοφορίες. Ε, αλλά η ώρα των ψηφοφοριών είναι στις 5. Οπότε έχουμε μισή ώρα διάλειμμα για καφέ ή ό,τι άλλο θέλετε. Συζητήσεις, κουβεντούλα και τα λοιπά. Ραντεβού στις 5 για τις ψηφοφορίες. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε νωρίτερα, διότι ο κόσμος έχει ειδοποιηθεί ότι ψηφίζουμε στις 5. The voting starts. So, uh, uh thank you all uh, so far. Σας ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ να επιστρέψετε στις 5 για να ψηφίσουμε. Λίγο πριν τις 5 προφανώς. Ευχαριστώ πολύ. Υπότιτλοι Are you ready to start the voting session? Είστε έτοιμοι για τις ψηφοφορίες. Um, the request for split vote. Για, τα, για τις χωριστές ψηφοφορίες ε, όσον αφορά τη συμβολή στον διερθρωμένο διάλογο έχουμε ε, λάβει δύο αιτήματα από το ΕΛΚ και από την ΚΟΕ για κατατμήματα τμήματα ψηφοφορίες ε, είναι ιδιαίτερες οι περιστάσεις. Θα επιτρέψω να γίνει κάτι τέτοιο σήμερα, αλλά πρόκειται περί εξαίρεσης και ε, είναι κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχε δεχθεί ο κανονικός πρόεδρος, γιατί κανονικά αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να συζητούνται στις συναντήσεις των σκιωδών και των συντονιστών προκειμένου να μην ε, μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά θα προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία, χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα. παραδεκτό των ε, ψηφοφοριών κατά τμήματα. Ολόκληρο το κείμενο χωρίς τα τα τμήματα 2 και 3. Θα γίνει ψηφοφορία επί ολόκληρου του κειμένου χωρίς τα τμήματα 2 και 3. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά.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 Those in favor. Ποιοι είναι υπέρ. Εντάξει, λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. First part, whole text without part two. Πρώτο τμήμα. Ολόκληρο το κείμενο, δηλαδή χωρίς τα τμήματα 2 και 3. Ψηφίσατε στα μηχανηματάκια σας. και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Χωριστή ψηφοφορία που ζητήθηκε από την ΚΟΥΕ. Στην παράγραφο 6 λοιπόν, η διατύπωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμίσου, Εξαμήνου και σε όλα τα στάδια του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Those in favor. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θεωρώ ότι απορρίπτεται. Όχι, ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. The vote is open. Έναρξη της ψηφοφορίας. The vote is closed. της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο τρίτο τμήμα, χωριστή ψηφοφορία που ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στην παράγραφο 8, η φράση «και προκειμένου να ενισχυθεί η νομοθεσία σχετικά με την άδεια πατρότητας υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει και εδώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. The vote is ψηφοφορίας εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. Προσθήκη 1. Πρόκειται για μια προσθήκη στην παράγραφο 6. Αν εγκριθεί, θα τοποθετηθεί στο τέλος του παραγράφου 6. Υπέρ, κατά, Αποχές, εγώ λέω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε βέβαιοι. Έναρξη vote open. ψηφοφορίας και πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προσθήκη νούμερο 2 που αφορά την παράγραφο 7. Αν εγκριθεί, θα τοποθετηθεί η προσθήκη αυτή στο τέλος της παραγράφου 7. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται λέω εγώ, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορίας παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία ε, σχετικά με τη συμβολή της Επιτροπής Απασχόλησης για τον διαρθρωμένο διάλογο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Και τώρα μπορούμε να επανέλθουμε σε μια πιο συνηθισμένη διαδικασία ψηφοφορίας. Περνάμε στην ψηφοφορία για την μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ και εισηγητής είναι ο κύριος ε, Πυρίνσκι. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 11, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Λοιπόν, απερίφθη. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός ε, Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ε, Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση από τη τροπολογία 23, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασα. Εγκρίνεται. Τροπολογία μάλλον όχι, συμβιβασμό C, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35, όχι συγγνώμη, συμβιβασμός D, υπέρ, κατά αποχέσε εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Θα την ψηφίσουμε. Τροπολογία 38 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχέσε, απορρίπτεται. Συμβιβασμός Ι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, όχι, καμία τροπολογία. Τροπολογία 51 διορθώνει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβασμός H στη σελίδα 9, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση επί της ε, συμβιβαστικής H, πέρα της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 67 και τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ, κατά, αποχέσε απορρίπτεται. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά, αποχέσε απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, ωραία, τροπολογία 70, ηλεκτρονική επαλήθευση, πέρασε της ψηφοφορίας Απερίφθη. Τροπολογία 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν επί του τροποποιημένου κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται 37 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Περνάμε λοιπόν στη, με την τροπολογία 74 για τους πρόσφυγες Μπράντο Benify. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι το 10 πριν από το 9 που ψηφίζουμε. Ε, η τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε για την 20, 82, συγγνώμη, παρακαλώ. η ψηφοφορία, η οποία και λίγη. Απορρίπτεται. τροπολογία παρ' 85 ψήφι υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 86 ε, κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές. Δεν ξέρω τι ψηφίζετε, οπότε το τσεκάρουμε αυτό ηλεκτρονικά. Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 86. Τελειώσαμε. 36 είπε Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, πάντα στην 86, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική. Ορίστε, θέλετε να το τσακάρουμε, παρακαλώ. Το δεύτερο τμήμα στην τροπολογία 86, ηλεκτρονική επαλήθευση, η οποία αρχίζει τώρα. Και τελειώνει κιόλα. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 91, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπέρ 100, υπέρ, κατά, Α, όχι, όχι, έχει κατά τμήματα, διορθώνει η Πρόεδρος. Το πρώτο τμήμα, λοιπόν, στην 100, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα το δεύτερο τμήμα της 100 υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον απορρίπτεται, αλλά θέλει έλεγχο. Εντάξει, ναι, θα το έλεγξω. Ηλεκτρονικά, λοιπόν, αρχίζει και κλείνει η ψηφοφορία. Ναι, έχει απορριφθεί. Όντως, η τροπολογία τώρα 102 και 103 μαζί ε, ε, ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική δέλτα D κατά αποχές. Τι γίνεται εδώ. Εγκρίνεται. Είναι τετρακανή, άρα εγκρίθηκε. Πού πάμε τώρα. Compromise DA. Συμβαστική DA. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία. 115 ψήφι υπέρ, Ε, ε, συγγνώμη, συμβαστική δεν την είδα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 115. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 120, το πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική F ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική H λέει η πρόεδρος, όχι έχει άλλες πριν. Την F πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα. 123, 124, 125 είναι ίδιες και ε, τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίφθεται Compromise H, η συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μητροπολογία 133, ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 149 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. Η συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Συμβαστική K, κάπα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές θα απορρίπτεται. Η συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 στη σελίδα 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ θέλετε για την 192. Άρχεται η ψηφοφορία. Και κλείνει κιόλα. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 195, 196 και 197. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβιβαστική π υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική Q καταπίπτει πώς καταπίπτει 203 έχει καταπέσει. Όχι, μια στιγμή. όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε. Καλά. 203 λοιπόν ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 216 έχει καταπέσει. Μια στιγμή να δούμε τι συμβαίνει είναι συμβατή λέει με τη 15, αλλά πρέπει να ψηφιστεί μαζί με την επόμενη. 216 and 217 are... 216 uh, και 217 είναι ταυτόσιμες και τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 και 225 ομού ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική S. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 234. Ε, υπέρ Όχι, 2.34. Γιατί εγκρίθηκε η υδροπολογία 133. Καταπίπτει η 2.31. Πάμε στην 2.34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ λέω ότι εγκρίνεται. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για την υδροπολογία 234, παρακαλώ. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Αναφέρεστε στην τροπολογία 234. Η ένστασή σα είναι για την τροπολογία 234. Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 234. Ωραία. Ας ξαναπάμε. Να ψηφίσουμε επί της τροπολογίας 234. Παρακαλώ ψηφίστε. Να ψηφίσουμε για την τροπολογία 234. Τέλος της ψηφοφορίας. Επί της τροπολογίας 2.34 και εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 235 και την ε, τροπολογία 236 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.37 υπέρ. Κατά το πρώτο τμήμα, συγγνώμη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 238. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εμένα μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε βέβαιοι. Επί της τροπολογίας 238, παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Συμβαστική SA υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 240 υπέρ, κατά, Α, εγκρίνεται. 242, 243 και 244 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 252 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική U παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DD. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2.59 και 2.60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 261. <clears throat> Καταπίπτει. Επειδή εγκρίθηκαν οι προηγούμενες δύο και πάμε στην τροπολογία 262 και 263 μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 264. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K. Ε, υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι πολύ σαφές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Συμβαστική KA. Παρακαλώ ψηφίστε. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.95 στη σελίδα 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 300 υπέρ, κατά, αποχές. Εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, όντως απορρίπτεται. Τροπολογία 302 υπέρ κατά αποχές εμένα μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Συμβαστική BB A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19, της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 306 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 307 μαζί με την 308 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Y υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Μπορεί και να κάνω λάθος. Ήταν λίγο ασαφές, πράγματι. Ας ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική Z. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 317 μαζί με την 318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 342 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 343 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 344 υπέρ κατά αποχές ε, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ τώρα Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική CC υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 364 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 365 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 367 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 374 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 376 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία προφορική των σοσιαλιστών 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία της Επιτροπής Πολιτισμού 23 συγγνώμη ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελογικές σκέψεις τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 Συγγνώμη, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά θα έλεγα. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Και όντως απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά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 Να ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπ... Ε, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Όχι. Συμβαστική ΙΙ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. FF, συμβαστική FF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός GG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία... Τι θέλετε? Ωραία. Ε, η ηλεκτρονική επαλήφωση για την τροπολογία 41 άρχεται η ψηφοφορία και ολοκληρώθηκε, έκλεισε μάλλον, και απερίφθη. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές τι να σας πω. Επαλήθευση. Τροπολογία 46. Άρχεται. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω ότι θα πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 50. Πέρας. Και απερίφθη όντως. Συμβιβασμός HH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε προφορική τροπολογία από τις τροπολογίες 60 που αφορά την διαγραφή της λέξεως adequate η οποία χρησιμοποιείται δύο φορές υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρο... Ε, συμβιβασμός JJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 και εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα ξεκινήσουμε την τελευταία ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Και η έκθεση εγκρίνεται λοιπόν με 36 ψήφους υπέρ και 8 εναντίον. E- λοιπόν, τώρα έχουμε σύμφωνα με τον κανονισμό συμπερίληψη τώρα των ψηφοφοριών στην έκθεση. Η κυρία Στέβενς παρευρίσκεται βεβαίως για να μπορέσουμε να αρχίσουμε και να ψηφίζουμε το σχέδιο αξίσχυα Στέβενς. Πέτη 6 της Επιτροπής Αναφορών. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέτη 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέτη 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φαμ 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άφετ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίβε 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 25 καταπίπτει. Όπως και η Τραν 8 και η Γιούρι 1. Άρα πάμε στη Βαστική 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα μάλλον είναι αυτή. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 20 ψήφιπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 46, έτσι δεν είναι, όχι. Πάμε στην επόμενη σελίδα, 47. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική L, ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική M υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος. 24. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. 24 της Επιτροπής Αναφορά. Πέρασε. Εγκρίνεται. ΕΝΒ 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται έλεγχος για την 60 Εγκρίνεται. 61. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Χρειάζεται πάλι έλεγχος για την 61. Αρχίζει. It is now closed and it's carried. Εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 63 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 64 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. Στην επόμενη σελίδα, συμβαστική πη ε, ε, λατινικό είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο, μάλιστα, για τη συμβαστική π, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε do we go to France? Compromise Q. Compromise Q. Oh, compromise Q on page 9. Those in favor. Q, ο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέ. κατά αποχές γκρίνεται. 83 υπέρ carried. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέ. κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τραν 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 7 χωριστή σε τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα And the vote is open. Αρχίζει ψηφοφορία. Closed. And it... Πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΕΡ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Amendment 88, those in favor, those... Uh... 8 υπέρ, κατά αποχές Μάλλον πρέπει να το ξαναψηφίσουμε γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Πολλές αποχές βλέπω. 88. Το 88. Γεμάτο αποχές είναι, καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Για να δούμε που θα καταλήξουμε πέρας. Αυτό είναι. It's carried. Εγκρίνεται, αλλά με πολλές αποχές. Ε, Γιούρι 10 πάμε τώρα. Είπε κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 90 υπέρ όχι καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η Γιούρι 10 πάμε στη Γιούρι 11 λοιπόν στη σελίδα 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ΤΑΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV20 nv 20 ειπε κατά ορίστε συγγνώμη Excuse me, chair. Sorry to... Ζητώ συγγνώμη, κυρία Στέβενς, που σας διακόπτω. Θέλω να επανέλθουμε στην τροπολογία 88. Είπατε ότι εγκρίθηκε, αλλά αν είναι περισσότερες οι αποχές από τα υπέρ, δεν ξέρω ε, κατά πόσο εγκρίνεται αυτή η τροπολογία. 29-28 ήταν οι αποχές. Ε, απήχαμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω αυτό να σημαίνει αυτόματα έγκριση με 12 υπέρ και 29 αποχές. Yes, but the expertise says that. Ναι, αλλά οι εμπειρογνώμονες μου λένε ότι δεν μετράνε οι εποχές. 12 υπέρ ήτανε ένας κατά και 29 αποχές. Άρα εγκρίνεται. Έτσι λένε οι ειδικοί. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μα 50% δεν πρέπει να υπερψηφίσουν των, τον ψηφισάντων. Ξέρω εγώ. I rely on... Uh, εγώ επαφίομαι στους ειδικού εδώ στην γραμματεία. Έτσι λένε οι κανόνες και οι κανονισμοί. Compromise T Συμβαστική τάφη μας ανεγρήθηκε και επανερχόμαστε που είχαμε μείνει. Στην MV20. Εγκρίθηκε και αυτή. Και τώρα πάμε... Α, όχι, πρέπει να ψηφίσουμε την MV20. Δεν είχαμε τελειώσει. Πάμε λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Σελίδα 15. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη είναι η 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. Η συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 544 υπέρ Κατά. Αποχέ carried. Αποχές εγκρίνεται. Φαμ 20 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 106 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Η συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107, 110 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική W, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία, όχι. Συμβαστική X, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 118. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 118 εγκρίνεται. Συμβιβαστική AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AB. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ...142 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί της 142. Παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Envy. Όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 144 υπέρ κατά αποχές εμένα μου φαίνεται ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί της 144 παρακαλώ ψηφίστε τώρα ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την 144 ναι εγκρίνεται λοιπόν 145. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AH υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 148 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Κουλτ. Ένα. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, τι θέλετε. Ωραία, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 148, παρακαλώ. Παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. Τέλος της φοφορίας. Εγκρίνεται. Κουλ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, κουλτ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, κουλτ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, κουλτ 9 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κουλτ 9. Ψηφίστε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία Και εγκρίνεται. <laughs> Με συγχωρείτε. Να, διαβάσ... να ψηφίσουμε για τις 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 μαζί, υπέρ. Εσείς λέτε όχι. Ωραία, ξεχωριστά. Κουλτ 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κουλτ 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κούλτ 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κούλτ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κούλτ 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέτη 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φά 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέτη 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV17 Υπε, κατά 8 εποχές εγκρίνεται, NV18 υπέρ κατά εποχες εγκρινεται εγκρίνεται, NV22 υπέρ κατά εποχες εγκρινεται εγκρίνεται, NV24 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται, NV25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται, NV26 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 9 υπέρ κατά αποχή. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ρέτζι 9. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, φαμ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, φαμ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, φαμ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, πέτη 50, όχι, ε, φαμ 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΦΑΜ 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 1 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. <clears throat> Τραν 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 3. Τραν 2 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Uh, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Τραν 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 10 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί της Τραν 10. Τραν 10, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τραν 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 12 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέτη 7, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέτη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Γιούρι 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Γιούρι 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Γιούρι 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Λίμπε 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Λίμπε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα λοιπόν, Λίμπε 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 27 υπέρ κατά α, αποχές. Λίμπε 27 ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε και εγκρίνεται. Λίμπε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 9 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. 9 ναι, πάντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την ΔΕΒΕ 20 άρχεται η ψηφοφορία και πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Αφετ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός AC υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 157 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Λίμπε 41 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 158 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 158. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. Πέτει ένα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 2. Καταπίπτει η Γιούρι Το ίδιο και η επόμενη. 159. Τροπολογία 159. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 160. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέτη 12. Υπέρ είναι στη σελίδα 32. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 161. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 163. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός AD. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός ΑΕ e. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 ε, καταπίπτει και περνάμε στο συμβασμό. Α, όχι, τη ψηφίζουμε την 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV30 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται ΦΑΜ 23 υπέρ... Α, όχι, καλύπτεται η ΦΑΜ 23. Συμβασμός ΕΙΕΦ υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 173 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πηγαίνουμε τώρα στο συμβιβασμό AG, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5-8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5-17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πέτει 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις, συμβιβασμός B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τραν E καταπίπτει. Είμαστε τραν A, τραν α, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τραν B, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός C, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός H, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία διαμαρτυρίες. Τροπολογία 12 ήταν πολύ σαφέ το αποτέλεσμα, λέει η πρόεδρο. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβιβασμό ή υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Φαμ, σι, φαμ, σι, υπέρ, κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Φαμ δι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε ει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ αι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ Ε υπέρ κατά J ε, και πηγαίνουμε μετά στην τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 28 29 και 30 μαζί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι η τροπολογία 33 θα πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 33 λοιπόν. Φαμ και όχι. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται λέτε εσείς. Καλύτερα να επαληθεύσουμε. Ε, έλεγχος λοιπόν ηλεκτρονικός από της τροπολογίας 34. Πέρα της ε, ψηφοφορίας. Ε, ναι, εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φαμ G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λέω εγώ, νομίζω. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα με την τελευταία ψηφοφορία ε, στο κείμενο έτσι όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία, είναι ηλεκτρονική, άρχεται η τελευταία αυτή ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασα 41 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι εναντίον. Το αποτέλεσμα αυτό θα ενσωματωθεί στην έκθεση και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Στίβενς ε, για την εργασία της. Ξέχασα όμως να συγχαρώ και τον κύριο Μπονιφάη προηγουμένως, ε, καθώς επίσης και τους ε, άλλους ε, εισηγητές. Η επόμενη συνεδρίαση είναι τη 15η Ιουνίου. Σας υπόσχομαι ότι στις 15 Ιουνίου δεν θα έχουμε τόσες πολλές ψηφοφορίες γιατί αυτό είναι πολύ σκληρή δουλειά. Σας ευχαριστώ πάντως για την συνεργασία.